όπου θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία.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 Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was.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 Πρόεδρος. Thank you. Uh, dear colleagues, please take... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. We'll begin in 30 seconds. Θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες σε μισό λεπτό.